σχέδιο Γενικού Προπολογισμού 2015 και σας ενημερώνω ότι δεν προβλέπεται διαδικασία Catch the για το θέμα αυτό, ούτε μπλε κάρτας. Επομένως μόνο οι συνάδελφοι που έχουν αγραφεί στον κατάλογο θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Και πριν καθυστερήσουμε περισσότερο θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσανέτσι εκ μέρους του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κύριε Επίτροπε, είναι τιμή για μας να βρίσκομαι εδώ και να σας παρουσιάσω τις θέσεις ε, του Συμβουλίου για το σχέδιο προπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, το οποίο εγκρίθηκε επισήμως τις 2 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για το νέο προπολογισμό στα πλαίσια του νέου ε, πολιετούς ε, προγράμματος 2014-2020 και ε, θα πρέπει να δούμε και την έναρξη των προγραμμάτων αλλά και την ολοκλήρωση των ε, προγραμματισμού 2007-2013 που είναι στη φάση ολοκλήρωσης. Αυτό ακριβώς ε, είναι και αυτό το οποίο έλαβε υπόψη το Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει τι ακριβώ θα προτείνει για τον προπολογισμό του 2015, συνειδητοποιώντα απολύτω ότι θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη ε, χρηματοοικονομική στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για του στόχου τη ανάπτυξη και τη απασχόληση και φυσικά και για την ολοκλήρωση τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Λαμβάνονται υπόψη βέβαια αυτοί οι στόχοι, αλλά λαμβάνονται υπόψη και το γεγονό ότι τα προγράμματα και ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίε θα πρέπει να γίνονται σε ένα πλαίσιο βιωσιμότητα και δημοσιονομική πειθαρχία με βάση όσα ε, ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη-μέλη για τον εθνικό τους προϋπολογισμό. Με όλα αυτά λοιπόν θεωρούμε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, προσαρμόζεται καταλήλως στις απαιτήσει ε, αυτές και προβλέπει ότι το Ευρωπα... η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτει τον απαραίτητο προπολογισμό για το 2015 προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει και για να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν νέες παρεμβάσεις σε διάφορες τοπίες ώστε να έχουμε υγιή εκτέλεση του προπολογισμού. Ε, κυρίως όσον αφορά τις ε, ε, αναλήψεις υποχρεώσεων για τα μέτρα ανάπτυξης και απασχόλησης, για να ξεκινήσουμε κυρίως με την απασχόληση των νέων, επιβεβαιώνει ότι είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι για αυτές τις προτεραιότητες, όπως προβλέπουν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης και 27ης Ιουνίου. Επίσης υπάρχουν πόροι για άλλους τομείς, τηλεοπικοινωνίες, ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, μετανάστευση και έρευνα και όλα αυτά έχουν προκύψει από την ιδιαίτερη προσοχή που έχει δώσει το Συμβούλιο και σε αυτές τις προτεραιότητες. Αυτό παρά το γεγονός ότι στην έγκριση της απόφασης του το Συμβούλιο έβαλε υπόψη ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξοικονόμηση σε κάποιες ε, τομείς ε, θεωρεί ότι μπορεί να κάνει εξοικονόμηση και θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν αρκετά περιθώρια για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τυχόν απρόβλεπτες ε, δαπάνες. Και επίσης ε, βασίσαμε τα πάντα σε μια εισβάθος ανάλυση των προγραμμάτων, κυρίως όσον αφορά τις βασικές ε, πραγματικές ανάγκες δαπανών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα απορρόφησης το 2015. Και επομένως φροντίσαμε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την έναρξη νέων προγραμμάτων, αλλά ούτε και για το κλείσιμο των ε, παρεμβάσεων οι οποίες είναι εξελίξη. Ε, η θέση του Συμβουλίου προβλέπει ένα προσωρινό προπολογισμό του 2015 που ακόμα και με αυτές τις μειώσεις που θεωρήθηκαν απαραίτητες και ε, θεωρήθηκε επίσης ότι είναι δυνατό να γίνουν προβλέπει αύξηση και για τις αναλήψεις υποχρεώσεων αλλά και για τις πληρωμές σε σχέση με τον προπολογισμό του 2014. Είναι δεδομένο βέβαια ότι το Ιταλία ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προπολογισμό του 2005 σε ένα επικοδομητικό πνεύμα και συνεργασία όπως πάντα γίνεται με τα τρία θεσμικά όργανα για την αναζήτηση συμβιβασμού για τον προπολογισμό. Να δούμε τώρα λίγο λεπτομερώς τη θέση του Συμβουλίου. Πρόκειται για μια θέση η οποία προβλέπει συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων 145 δισεκατομμυρίων ευρώ και 140 δισεκατομμύρια ευρώ για τις πληρωμές. Όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπεται μία μείωση 522 ε, εκατομμυρίων ευρώ για τις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων και 2,2 δισεκατομμυρίων για τις πληρωμές. Όπως σα είπα ήδη, παρά το γεγονό ότι υπάρχουν αυτές οι μειώσεις και στις αναλήψεις υποχρεώσεων και στις ε, πληρωμές υπάρχει αύξηση του προπολογισμού σε σχέση με το 2014, λαμβάνοντας υπόψη και τον ε, διορθωτικό προπολογισμό του 2014 που έγινε. Υπάρχει 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, ε, είμαστε λοιπόν στο 1,75% και αύξηση τη τάξη των 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που σημαίνει ότι είμαστε στο 3,32% ε, αύξηση. Και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να επισημάνουμε λοιπόν ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν προβλέπει καμία ε, προσαρμογή του, ε, του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε σύγκριση με το 2014 και σε σχέση με τα ο διορθωτικούς προπολογισμό του 2014 που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τους οποίους ακόμα κάνει αξιολόγηση το Συμβούλιο. Γι' αυτό ακριβώς, όπως επιβεβαίωσα και προηγουμένως, πρόκειται για μια θέση η οποία εξισορροπεί τις ανάγκες κατάλληλη προσαρμογής τη πολιτική ε, κοινοοικονομική ανάπτυξη που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανάγκη ταυτόχρονα βιωσιμότητα και πειθαρχία του προπολογισμού. Πολλό δε μάλλον να λάβουμε υπόψη και την δήλωση ε, της θέσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από την οποία ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προταθεί διορθωτικός ε, προϋπολογισμός, αφή στιγμή ε, οι αναλήψεις υποχρεώσεων και οι πληρωμές του 2015 θεωρηθούν ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ε, κυρίως για τους τομείς στους οποίους υπάρχουν υπόλοιπα προς εκαθάριση το θέμα αυτό στο Συμβούλιο καταλήξαμε σε μια ευρύτατη συνένεση και υπάρχει σχεδόν πλήρης αποδοχή από όλα τα κράτη-μέλη. Και τώρα δεν θα ήθελα να ε, μπω σε λεπτομέρεια σε κάθε θέμα, ε, αλλά είμαι στη διάθεσή σας βέβαια ε, στη συνέχεια για περαιτέρω διευκρινήσεις, αλλά να επαναλάβω ότι και για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού την οποία η θέση ε, του Συμβουλίου είναι πάντα ε, μία μικρή αύξηση ε, σε σχέση με τον προπολογισμό του 2014. Να σας πω συνοπτικό ποιες είναι οι τρεις αρχές οι οποίες ε, ε, αποτέλεσαν το νήμα της σκέψης ε, του Συμβουλίου για το προπολογισμό του 2015. Καταρχάς, η ανάγκη να προβλέψουμε κατάλληλη πρικοδότηση για τις πολιτικές οι οποίες ενδιαφέρουν περισσότερο τους Ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή την καταπολέμηση της ανεργίας, κυρίως της ανεργίας των νέων, επενδύσει στην έρευνα και στην καινοτομία, υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαχείριση των διεθνών κρίσεων, όπως για παράδειγμα της κρίσης της Ουκρανίας και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και ανθρωπιστική βοήθεια. Δεύτερον, η ανάγκη να επαγρυπνούμε για τα δημόσια οικονομικά, λαμβάνοντα υπόψη και τι σημαντικέ προσπάθειε που ζητούνται από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να συγκρατήσουν του προπολογισμού του. Κυρίω θα πρέπει να προσέξουμε να ελέγξουμε τι διοικητικέ δαπάνε ε, και να πούμε ότι εμεί εμπιστευόμαστε τη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Διοίκηση να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο να διαχειριστεί του πόρου του. Και τέλο, η ανάγκη να υπάρχει ένα λογικό προπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάτω από τα μέγιστα όρια τα οποία προβλέπονται για τον ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα όσα ε, χρειάζονται. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η θέση της του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θεωρείται από την Ιταλική Προεδρία ότι είναι μια ισορροπημένη θέση ε, η οποία κάνει κατάλληλη διαχείριση των πόρων για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ταυτόχρονα με την ανάγκη της εξυγίασης των δημοσίων οικονομικών, η οποία ανάγκη αφορά και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο των κρατών μελών. Επίσης, να σας πω ότι η Ιταλία θα συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να βρούμε ένα συμβιβασμό για τον προπολογισμό του 2015, που να λαμβάνει υπόψη και τις ευαισθησίες και τις προτεραιότητες των τριών θεσμικών οργάνων. Ολοκληρώνοντας, να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει μια επικοδομητική ε, και ε, σωστή αντιπαράθεση και είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και στοιχεία. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Zanetti. I'll now give the floor. Ευχαριστώ κύριε Τσανέτη και τώρα παρακαλώ τον κύριο Ντομινίκη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Υπουργή. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ σε εσά σήμερα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια της ε, Προεδρίας ε, ε, για τον σημερινό και τους επόμενους προπολογισμού. Δύο νούμερα θέλω να σας δώσω. Το, το προπολογισμό του 2014 αν υιοθετηθεί με όλες τις τροπολογίες που έχει προτείνει η Κομισιόν, θα εξακολουθήσει να είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου κάτω από τις ε, πληρωμές του 2013. Ενώ ο προπολογισμό για το 2015, αν υιοθετηθεί όπως τον προτείναμε, και πάλι θα είναι ακόμα 2 δισεκατομμύρια χαμηλότερος από τον προϋπολογισμό του 2013. Οπότε ε, είμαστε πολύ μακριά από τις παλαιότερες, από τα παλαιότερα ύψη δαπανών στα οποία ήμασταν συνηθισμένοι. Υπάρχει μια αύξηση του προπολογισμού το 2015 λέχθηκε, όμως στην πραγματικότητα τα ποσά μειώνονται αν τα μελετήσετε προσεκτικά. Τώρα, πρέπει να πω ότι σήμερα η Κομισιόν θα πρέπει να επαναλάβει την ε, θέση της, είναι απογοητευμένη από την ανάγνωση του Συμβουλίου για το προσχέδιο Προπολισμού του 2015. Το Συμβούλιο ε, ε, δεν παρακολουθεί την, την πρωτοφανή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η Κομισιόν έχει ε, μελετήσει την κατάσταση στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της διαδικασίας, της δημοσιονομικής διαδικασίας, θέλω να προστιαστώ στα εξής. Η πρόταση της Κομισιόν για τον Προπολισμό του 2015 ε, συντάχθηκε σε μια περίπλοκη δύσκολη συγκύρια. Ε, ο βασικός μας ε, στόχος είναι η, καταρχήν η οικονομική ανάπτυξη με προγράμματα που θα δώσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και ε, θέσεις εργασίας ε, στόχους στόχοι οποίοι είναι και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. θα πρέπει η μεγαλύτερη δυσκολία όμως αφορά τις πληρωμές. Πρώτον, θα πρέπει να έχουμε επαρκή κονδύλια για την χρηματοδότηση των πολιτικών προτεραιοτήτων, τις οποίες ε, συμφωνήσαμε στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεύτερον, θα πρέπει να βρούμε μια λύση και να ελέγξουμε τις ε, κρεμούσες πληρωμές, να πληρώσουμε τα ε, τιμολόγια ε, της περίοδου 2007-2013 που εκκρεμούν και να επιστρέψουμε δαπάνες στα κράτη-μέλη και σε άλλους δικαιούχους σε ένα λογικό χρονικό περιθώριο διάστημα. Για να το πετύχουμε αυτό, η Κομισιόν πρότεινε να χρησιμοποιήσει όσους πόρους έχουμε το 2015 και την μέγιστη δυνατή ευελιξία που προβλέπεται από τις σημερινές δημοσιονομικές προοπτικές. Σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες, η Κομισιόν πρότεινε ε, την αύξηση κατά 5,8% στις ε, αναλήψεις πληρωμών και ανάληψη σχεδόν 13% στις πληρωμές. Αυτό χρειάζεται για να καλυφθούν τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο επέστρεψε στην παραδοσιακή του τάση να μειώνει τι ε, για κατά μισό δισεκατομμύριο ευρώ και τις πληρωμές κατά πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Με πάνω από το 60% περικοπών να ε, ε, αφορούν τον ε, τίτλο 1α, που είναι ο τίτλος το, που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για του νέου. Για το τίτλο 1α οι ε, περικοπές ε, φτάνουν στο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πληρωμές. Για την έρευνα η μείωση 10% η οποία θα επηρεάσει το ορίζον 2020 ε, και 600 ερευνητικά προγράμματα με 7.000 περίπου συμμετέχοντες. 140.000 από αυτούς είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, επίσης, εξωτερική πολιτική. Παρόλη την ε, δέσμευσή μας να είμαστε δραστήριοι και ενεργοί, ιδιαίτερα με τις γειτονικέ χώρες, οι σημαντικές ε, μειώσεις κατά 344 ε, εκατομμύρια ευρώ προβλέπεται από το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε όλες τις πληρωμές που μπορούμε να διαθέσουμε, που προτείναμε και για το 2014 και για το 2015 και να χρησιμοποιήσουμε πλήρω την αρχή τη ευελιξία αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, όρια στην μετάθεση πληρωμών για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι ε, αυτό που ζήτησε η Κομισιόν το 2015 μπορεί να επαρκέσει μόνο ε, αν κάνουμε ότι πρέπει το 2014. ο ετήσιος προπολογισμό μα εφαρμόζει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν αλλάζει την πολιτική συμφωνία. Οι πολιτικές ε, συμφωνίες έγιναν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα τις εφαρμόζουμε μέσω των ετήσιων προπολογισμών. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση ε, που, όπου το 2014 δεν είχαμε παρκή κοντιλέ για τις πληρωμές, η Κομισιόν λυπάται για τη θέση του Συμβουλίου στην ανάγνωση του προπολογισμού 2015. Το Συμβούλιο δρά ε, σαν να μην υπάρχει κάποια έκτακτη κατάσταση, αγνοώντας ε, τις προτεραιότητες και την κατάσταση του προπολογισμού. Η, αυτή η προσέγγιση δύο σταδίων ε, με, μια, ένα χαμηλό επίπεδο πληρωμών και ένα ενδεχόμενο πρόσθετο προπολογισμό και διάρκεια του έτους δεν είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Γιατί δημιουργεί προβλήματα ρευστότητα στον ετήσιο προπολογισμό. Σα κάνω έκκληση, εσά προ το Κοινοβούλιο, να λάβετε υπόψη αυτέ τι ανησυχίε στην προετοιμασία τη δική σα ανάγνωση του προπολογισμού το 2015. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να ε, σπάσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο με την ε, ε αναβολή των πληρωμών. Για να υλοποιήσουμε τις κοινέ μας ε, προτεραιότητες, ε, να ε, φέρουμε σε πέρα τις υποχρεώσεις μας σε ό,τι αφορά τις αναλήψεις τις πιστώσης αναλήψεων υποχρεώσεων. Οι προτάσεις πληρωμών για το 2015 από πλευράς της Κομισιόν θα βοηθήσουν έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του 2014, στις πληρωμές του 2014, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πληρωμές ε, θα ληφθούν υπόψη στον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 3 για το 2014 με την ε, έκκληση να χρησιμοποιηθεί ε, το υπολοιπόμενο ε, περιθώριο των 700 εκατομμυρίων ευρώ και η εξελίξη ό,τι αφορά τις, ε, ε, τα έσοδα θα πρέπει επίσης να κινηθούν προς την, αθή, προς την διακατεύθυνση. Αν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα, τότε ε, οι πληρωμές του 2014 θα γίνουν χωρικός κόστος για τα κράτη-μέρη. Αυτό σε μια περίοδο στενών εθνικών προπολογισμών θα πρέπει να υποφελθούμε τη ευκαιρία για να ελέγξουμε και να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Τέλος πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη την ευελιξία που προβλέπεται από το καινούριο δημοσιονομικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτες καταστάσεις και για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση των πληρωμών. Ε, περιμένω με ανυπομονησία την ε, συνάντησή μας 24 Σεπτεμβρίου για να βρούμε ε, μια βιώσιμη προσέγγιση. Θα ήθελα ήδη να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την ε, πρωτοβουλία του ε, ε, να συγκαλέσει αυτή την διοργανική διάσκεψη και ιδιαίτερα τον κύριο Αρτουά, πρόεδρο της Επιτροπή Προπολισμών και τον εισηγητή για το 2014 και 2015, την εισηγήτρια, κύριε ε, Χόλχερμαρ, τον κύριο Ντεπρέ και την κυρία Ίδια Θάβαλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο και τώρα δίνω το λόγο στους, στις δύο συνεισηγήτρες, την κυρία Χολμάιερ πρώτα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλωσορίζω και την Προεδρία. Θα ήθελα καταρχάς αγαπητοί συνάδελφοι να επισημάνω παρότι είμαι αρμόδια εκ μέρους του Κοινοβουλίου για τα λοιπά τμήματα να πω προς την Επιτροπή ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνομαι πλέον τι κάνει το Συμβούλιο. Έχουμε εγκρίνει ένα επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο φαίνεται ότι αγνοεί, δεν γνωρίζει πλέον τι περιλαμβάνει το Συμβούλιο. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Δεύτερον, έχουμε να επισημάνουμε ότι θέλουμε να ε, ενισχύσουμε τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη. Γιατί λοιπόν να περικόπτουμε ακριβώς τα συγκεκριμένα κεφάλαια, τα ποσά που προβλέπονται για την έρευνα και την τεχνολογία ή για τις θέσεις εργασίας. Όταν μιλούμε για ανθρωπιστική ενίσχυση προς τη Συρία και τις περιοχές κρίσεως, γιατί περικόπτεται τα σχετικά κεφάλαια στον προπολογισμό. Η ανάπτυξη που θέλουμε να ενισχύσουμε, γιατί να περικόπτονται τα σχετικά τη κεφάλαια. Πρέπει να πω επίσης ότι ύστερα από πολλέ διαπραγματεύσει που παρακολούθησα για του προπολογισμού, ανά τα έτη, βλέπω ότι δεν υπάρχει αντιστοίχηση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Πρέπει να έχουμε επαρκή ποσά για να τιμούμε τι υποχρεώσει μα και να καταβάλουμε τι πληρωμές. Φαίνεται λοιπόν σιγά σιγά το Συμβούλιο να έχει αρχίσει να διαχωρίζει τα λόγια από τα έργα του και δεν καταλαβαίνω πλέον όταν μιλούμε για ανάπτυξη και γνωρίζουμε και βλέπουμε ότι περικόπτονται τα κονδύλια για την έρευνα πώς είναι δυνατό το Συμβούλιο ενώ έχει το ίδιο δώσει τις σχετικές δεσμεύσεις για ανάπτυξη να προχωρήσει σε περικοπές. Εμείς έχουμε ως Κοινοβούλιο επιλέξει χωρίς ε, γενικές αυξήσεις να δώσουμε το βάρος σε άλλα σημεία του προϋπολογισμού. Έχουμε ε, ένα θέμα που έχει να κάνει με το καθεστώς των βουλευτών με διψήφιο ποσό περικοπών και εξοικονόμηση σπόρων και συνεχίζουμε με μια γραμμή λογική και ε, προσεκτική στις δαπάνες για την υπηρεσία εξωτερικής δράσεως ε, θα ήθελα να πω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη αλλά δεν έχει επαρκείς πόρους για να μπορέσει να αναλάβει δράση και να ε, επιτελέσει το έργο της κατά τρόπο ορατό. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, επαρκή ε, χρηματοδότηση ώστε να έχουμε επικοινωνία, ώστε να έχουμε γνώση της δράσης αυτής της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, ώστε να μην χρειάζεται μέσω του YouTube να μαθαίνουμε τι, έχουν δηλώσει, ε, τι έχει δηλώσει το προσωπικό της. Το ίδιο και για το δικαστήριο, διότι θα ήθελα να επισημάνω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε να κάνουμε με προσφυγές σχετικές με την βραδύτητα των οικονομικών διαδικασιών και ίσως τελικά θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι νέες θέσεις δικαστών για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε να μπορέσει να καλύψει το την πολύ σημαντική καθυστέρηση στις δίκες. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Τώρα η κυρία Γκάρδια Σαμπάλ Μπογιάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Τζανέτη, πίτροπε Ντομινίκ, ε, εκπλήσει ε, η σύγκληση των προτεραιοτήτων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και το πόσο μακριά βρίσκονται τελικά οι θέσεις σε σχέση με τον προπολογισμό. Μοιραζόμαστε προτεραιότητες αλλά όχι και θέσεις για τον προπολογισμό. Όπως είπα ε, και η Κομισιόν, μια σημαντική προτεραιότητα των οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βγούμε από την κρίση, ε, να δημιουργήσουμε ανάκαμψη, θέσει εργασία και να καταπολεμήσουμε την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων. Αυτά είναι μέτρα βραχυπρόθεσμα και πιο μακροπρόθεσμα μπορούμε να μιλήσουμε για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και ε, την επιτυχία του στόχου τη αύξηση τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο μα. Γι' αυτό το λόγο χρειάζονται επενδύσει. Πρέπει να επενδύσουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στον κόσμο της γνώσης. Ε, και θα πρέπει να ενισχυθούν τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη, την παιδεία, ε, βοήθεια ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και υποδομές και ενέργεια που είναι μια από τις σημαντικές προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Όμως όταν φτάνουμε στις λεπτομέρειες, όταν φτάνουμε στο πρακτέο ε, συγκεκριμένα κονδύλια κλπ. Διαφέρουν πάρα πολύ οι απόψει μεταξύ ε, ημών και του Συμβουλίου. Διότι εμεί στην ανάγνωσή μα και θα δείτε τη συμφωνία στην οποία θα φτάξουμε τι επόμενε μέρε θα ενισχύσουμε πολύ, πολλά από αυτά τα προγράμματα. Αντίθετα, εσεί στη δική σα ανάγνωση, το Συμβούλιο εννοώ εσείς, ε, περικόπτεται 198 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα, 35 εκατομμύρια στο μηχανισμό της Ευρώπη ε, ή 75 εκατομμύρια στα προγράμματα ε, ε, υποδομών μεγάλης κλίμακος. Υπάρχει λοιπόν μια αντίφαση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίζει το Συμβούλιο, τα Συμβούλια, το ΕΚΟΦΗΝ και όλα τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, όπως για παράδειγμα αυτό του, του Ιουνίου του περασμένου έτους και, τελικά, και, και αυτό που ε, τελικά πράττει το Συμβούλιο. Αυτά για την ανάληψη υποχρεώσεων. Για τι πιστώσει πληρωμών είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Με τη δική σα ανάγνωση του προπολογισμού, όχι μόνο δεν λύνεται τα προβλήματα, αλλά τα επιδεινώνεται. Τελειώσαμε το 2013 με 25 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, κρεμούσε πληρωμέ. Και αντί να αυξηθεί ε, ε, αυτή η γραμμή του προπολογισμού τιμιώνεται κατά 2,1 δισεκατομμύρια ακόμα. Δεν είναι επιβεβαιώσιμο αυτό ο προπολογισμό. Δεν θα μπω στη, σε τεχνικέ λεπτομέρειε. Η Κομισιόν μα εξήγησε. Να σα πω όμω δύο πράγματα. Πρώτον, η, η περικοπή του προπολογισμού των πληρωμών δεν ισοδυναμεί με εξοικονόμηση κονδυλίων. Το μόνο που κάνουμε είναι να μην πληρώνουμε αυτά που χρωστάμε. Ε, δεν τηρούμε τις συμφωνίες του δημοσιονομικού πλαισίου με αυτόν τον τρόπο. Το μόνο που κάνουμε ε, είναι να αναβάλουμε πιστώσεις οι οποίες είναι πολύ σημα... Ε, ζωτική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι διπλό το λάθος. Γιατί, γιατί αν πιστεύετε ότι θα λυθούν έτσι τα εθνικά οικονομικά προβλήματα με περικοπές από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, σίγουρα δεν θα το πετύχετε. Μακάρι με μια μικρή περικοπή του ευρωπαϊκού προπολογισμού να λύναμε τα προβλήματα των εθνικών προπολογισμών δεν αναγνωρίζουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό όραμα ως τέτοιο. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ιταλική Προεδρία να προσέξει πολύ προσεκτικά και από κοντά το θέμα των πληρωμών και να μελετήσει τις εναλλακτικές δυνατότητες λύσης του προβλήματος μέσα στο Συμβούλιο. Αν το αντιμετωπίσετε στην πράξη, το Κοινοβούλιο θα σας βοηθήσει και θα συνεργαστεί μαζί σας πολύ στενά. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκαμπριέλ Σαβάλ. Γκαρτία Ο κύριος Αχτφίμε τώρα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους Επιτροπή ε, των Προπολογισμών. Θα ήθελα να σα επισημάνω ότι έδωσαν πολύ αυστηρή ετοιμιγορία οι εκλογές του Μαΐου και είδατε με πόσο ισχυρούς ανέμους έπνευσε το πνεύμα του, ε, το αντιευρωπαϊκό ανησυχητικά επίπεδα δεν βλέπουμε στους νέους και ενώ το αντιευρωπαϊκό πνεύμα ε, μένεται ανά την ε, Ευρώπη το Διεθνές Νομισματικό Τομείο ανησυχεί για τη στασιμότητα στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν μπορεί η Ευρώπη να αποκαταστήσει τα προβλήματα και να εξασφαλίσει νέα εμπιστοσύνη. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τρει προποθέσει. Πρώτον, πρέπει να προετοιμάσουμε την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που υιοθετήθηκε το στα τέλη του 2013, το οποίο για 7 έτη ορίζει το ανώτατο όριο των δαπανών και το επίπεδο των εσόδων. Δεν μπόρεσε αυτή αυτό το πλαίσιο το οποίο θετέθηκε πριν από τις εκλογές να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των ψηφοφόρων. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη δυνατότητα να ε, χαλαρώσουμε έναν προϋπολογισμό από το 2015 και μετά, έναν ε, προϋπολογισμό αγωνιστικό δεδομένων των συνθήκων που αντιμετωπίζουμε. Ε, έχει νόημα να κλειστούμε σε μια δημοσιονομική σύραγγα στενή η οποία θα μας φέρει αντιμέτωπους με οποιοδήποτε ατύχημα θα βρούμε μπροστά μας. Έχουμε να κάνουμε με διαδικασίες που ξεκίνησαν το 2012-2013. Η Ευρώπη βρίσκεται ε, πρώτων θυρών μιας οικονομικής κατάρρευσης και αυτός ο προπολογισμό στον οποίο αναφέρεστε αποτελεί ε, σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια διαφορετική θεώρηση από τον προπολογισμό 2015 με ειδικέ ε, επιλογές και μέγιστες ε, επιλογές. Επίση, η απόκληση μεταξύ των δεσμεύσεων υποχρεώσεων και πληρωμών. Το Δεκέμβριο του 2013 είχαμε υπόλοιπα προς ρευστοποίηση όλο και μεγαλύτερα. Με 5 δισεκατομμύρια στα τέλη του 2010 είχαν γίνει 24 στα τέλη του 2013, αλλά απαγορεύεται από τι συνθήκε ε, η χρέωση τη Ευρώπη. Δεν μπορεί να αναλαμβάνει χρέο δηλαδή η Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι επιβάλλεται αυτή η πολιτική, η ύπουλη, αυτή η οποία θέτει σε κίνδυνο του ε, εταίρου ε, για ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με 1% μόνο, αντιστοιχούν στο 1% μόνο του ΑΕΠ της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει να βρούμε μια λύση συνετή, μια λύση όμως και συνεπή για να μπορέσουμε να εκαθαρίσουμε τα βάρη του παρελθόντος και να προχωρήσουμε με θετικά βήματα. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τα 300 δισεκατομμύρια των επενδύσεων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Επιτροπή τον ε, Ιούλιο εφέτος, από πού θα βρεθούν. Μόνο ε, όταν υπήρχε δυνατότητα χρηματοδότηση από τις αγορές ε, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αυτά τα ποσά. Η Ευρώπη όμως θα πρέπει να αναλάβει κίνδυνο εφόσον θέλει να μεγαλουργήσει και αυτό ο κίνδυνο σημαίνει ταυτόχρονα έκφραση στον προϋπολογισμό. Γιατί βλέπουμε όλοι πόσο κατεπίγουσα είναι η ανάγκη να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν θέλω με ιδιαίτερη έμφαση να υπογραμμίσω ότι ο προπολογισμό του 2015 δεν πρέπει να είναι μια απλή συνέχεια των προηγούμενων προπολογισμών. Δηλαδή να δίνει ακόμα ε, να συμπιέζει ακόμη περισσότερο τις δεσμεύσεις πληρωμών. Η Ευρώπη έχει ιδρυθεί, εμείς έχουμε εκλεγεί για να της δώσουμε νέα όθηση και πρέπει να τιμήσουμε την ψήφο των ε, πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να απαντήσει τώρα το Συμβούλιο στις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων και τα σχόλια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα ε, για μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση ανάλογα με τις ε, μακροοικονομικές εξελίξεις. Βέβαια, εδώ δεν θα πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Εδώ τώρα πρέπει να συζητήσουμε το σχέδιο προπολογισμού του 2015 δεδομένου του παρόντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι μπορώ να σας πω ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε τις προτεραιότητες. Αλλά σαφώς στις επιλογές εφαρμογής του, εκτέλεσης του προϋπολογισμού ακολουθούμε μία ε, σταδιακή προσέγγιση η οποία ξεκινά από την προϋπόθεση ή μάλλον ε, ξεκινά από δύο θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Πρώτον, όπως σας είπα προηγουμένως, μια θέση του ε, Συμβουλίου που οδηγεί σε ε, μεγαλύτερο προϋπολογισμό για το 2015 σε σχέση με το 2014 και σε καμία περίπτωση δεν είναι κατώτερος από αυτόν ο οποίος θα προέκυπτε εάν λαμβάναμε υπόψη και τις προτάσεις διορθωτικού προϋπολογισμού του 2014 που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρουμε ότι ακόμα αξιολογείται η θέση του Συμβουλίου. Αλλά για το 2015 η θέση του Συμβουλίου ήδη είναι ένα σημείο εκκίνωσης που σε σχέση με το προηγούμενο έτος ε, θεωρείται ε, καλύτερη. Δεν γίνεται καμία ε, προσαρμογή Και υπάρχει και η σχετική δήλωση του Συμβουλίου, η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει για το 2015 ε, διορθωτικό προπολογισμό σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητος ο διορθωτικός ε, προπολογισμό σε σχέση πάντα με τις πληρωμές όσον αφορά το θέμα της ανταγωνιστικότητας, τη ανάπτυξη και τη απασχόλησης, δηλαδή τη, ε, ε, σημείο 1α, θα ήθελα να σα ε, υπενθυμίσω λίγο τα αριθμητικά στοιχεία, διότι η θέση του Συμβουλίου εδώ είναι αναλήψεις υποχρεώσεων 17 ε, δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, σε μείωση 324 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αύξηση κατά 640 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2014 και οι πληρωμές είναι 14,2 δις ευρώ, με μείωση σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της τάξης του 1,3 ε, του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ, με αύξηση όμως σε σχέση με τον προπολογισμό του 2014 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει καμία μείωση σε σχέση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο κεφάλαιο αυτό από πλευράς ε, Συμβουλίου για τους πόρους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία μέσω του προγράμματος COSME, καθώς επίσης και για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων μέσω του προγράμματος Erasmus ΣΥΝ. Πρόκειται λοιπόν πληρωμές και για τον ορίζοντα 2020 και για τους μηχανισμούς για να ε, βοηθήσουμε την Ευρώπη. Ε, προτάθηκαν ε, και από το Συμβούλιο κάποιες μειώσεις μεν, αλλά έχουμε αύξηση σε σχέση με τον προπολογισμό του 2014. Ε, έχουμε μια αύξηση στο πρόγραμμα ΣΕΦ κατά 60% και το ορίζοντας 2020 22,3%. Το Συμβούλιο λοιπόν συνειδητοποιεί απολύτω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα συνεισφέρει ιδιαίτερα στην ε, ανάπτυξη και στην ε, απασχόληση, κυρίως δεδομένου ότι ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εξέλθουμε από μια παρατεταμένη χρήση. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε συγκεκριμένε προτάσει για τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω όσον αφορά την ενεργεία των νέων, την ε, χρηματοδότηση τη έρευνα και τη ε, καινοτομία και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά όπω υπενθυμίσαμε, το Συμβούλιο θα πρέπει ταυτόχρονα να επιδεικνύει και κάποιο ρεαλισμό, ο οποίο θα βασίζεται και στα ποσοστά χρήση των κονδυλίων στο παρελθόν, ε, και ε, ως προς τη δυνατότητα απορρόφησης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ βεβαίως για αυτή την ε, πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και είμαι βέβαιος ότι αν αντιληφθούμε ο ένας στη θέση του άλλου, θα έχουμε και την απαραίτητη προϋπόθεση για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2015 και θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση αποτελεί ένα πολύ καλό εφαλτήριο από πλευρά Ιταλική Προεδρία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμό με επικοδομητικό πνεύμα για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα στι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών, διότι γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα προπολογισμό ο οποίο θα ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των πολιτών και είμαι βέβαιο ότι ε, από κοινού το ε, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρουν τον κατάλληλο τρόπο για να αντιμετωπίσουν αυτό το στόχο. Ευχαριστούμε κύριε Τζανέτη. Με αυτό ολοκληρώνω τη συζήτηση για το σχέδιο προπολογισμού για το 2015. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι μια δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δομικές ελλείψεις όσον αφορά τις πληρωμές στον προπολογισμό του προγράμματος Horizon 2020 και να δώσω και πάλι το λόγο στο Συμβούλιο ε, στον κύριο Τζανέτη για να ξεκινήσει η συζήτηση. Θα σας αφήνουμε να πάρετε και μια ανάση.